και την αναγνώρισή μας προς τους άνδρες και τις γυναίκες που αφιερώνουν τις γνώσεις τους, το χρόνο και τη ζωή τους μερικές φορές ε, στην βοήθεια των συνανθρώπων τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, και για τις αντιδράσεις. Έχουμε 50 περίπου ψηφοφορίες ενώπιόν μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν να τις διεξαγάγουμε απρόσκοπτα. Η πρώτη έκθεση είναι της κυρίας Χάουταλα και αφορά την ε,